διάταξη. Η μερίσα διάταξη που εγκρίθηκε από το διάσκεψη των Προέδρων σας έχει διανεμηθεί. Στην ημερήσια διάταξη λοιπόν έχουμε καθορίσει τα εξή. Μετά από διαβουλεύσεις με τις πολιτικές ομάδες θα ήθελα να επιβάλλω την εξή αλλαγή για το οριστικό σχέδιο ημερήσια διάταξη. Η συζήτηση για το Σουδάν, περιπτώσεις Χασάν Αντουραχέμ και Αμπτουλομνέμ Αμπτουμαβάλα αντικαρθίσατε από τη συζήτηση για τη Ζιμπάμπουα την υπόθεση του ε, πάστορα Εύαν Μαβαρίρε. Υπάρχουν ενστάσεις. Εγκρίνεται λοιπόν η αλλαγή αυτή στην ημερήσια διάταξη. Για τη Δευτέρα, η ομάδα Ευρώπη των Εθνών και της Ελευθερίας ζήτησε η δήλωση της Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής υπάτου εκπροσώπου για την εξωτερικές υποθέσεις και την πολιτικές ασφαλεία για τις αποκαλύψεις Wikileaks για τη CIA ε, να ε, βρεθεί στο πρώτο σημείο στην ημερήσια διάταξη. Και έτσι η Ολομέλεια θα παραταθεί μέχρι τις 12. Να δώσω το λόγο στον κύριο Πρέτσελ για να παρουσιάσει το αίτημα του ΕΝΕΦ. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, ο Wikileaks δημοσίευσε τα πρώτα έγγραφα και λέει ότι θα αποδεσμεύσει και άλλα για τις δραστηριότητες της CIA που παρακολουθεί έξυπνα τηλέφωνα, ακόμα και έξυπνες τηλεοράσεις, μέχρι και αυτοκίνητα. Οι ΙΗ αυτοί μπορούν μάλιστα να τηλεκατευθύνουν υποσυνθήκες και αυτοκίνητα και βεβαίω η τεχνολογία αυτή σβήνει τα ίχνη της και δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι θα μπορούσαν ακόμα να τα χρησιμοποιήσουν αυτά οι πάλι CIA χωρίς γνώση καν της υπηρεσίας αυτής και μπορούν βεβαίω να σφύνουν ε, τα δικά τους ίχνη και να αφήνουν άλλα ε, υπότιθεται των ε, Ρώσων. Και έτσι βλέπουμε τα γεγονότα χάρη, της Γαλλίας το 2010 υπό διαφορετικό φως. Οι hacker της CIA έχουν ως βάση το προξενείο των ΙΠΑ στην Φραγκφούρτη για Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Αφρική. Η γερμανική κυβέρνηση μέχρι στιγμής αρνείται να τοποθετηθεί δημοσίως και απαιτείται να γίνει αυτή η συζήτηση όχι μόνο στην Γερμανία θεωρώ ότι είναι μια συζήτηση που αφορά όλες τις ευρωπαϊκές χώρες και θα πρέπει να γίνει εντός της αίθουσας αυτής σήμερα. Σας ευχαριστώ. Υπάρχει κάποιος ο οποίος θα ήθελε να παρέμβει κατά της πρότασης. Δεν θέλει κανείς να παρέμβει κατά. Ψηφίζουμε λοιπόν το αίτημα της Ομάδας Ευρώπη των Εθνών και της Ελευθερίας για να προσθέσουμε μια δήλωση της Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής υπάτης εκπροσώπου εξωτερικών υποθέσεων και πολιτικής ασφαλείας για τις αποκαλύψεις του Wikileaks για τις ε, μεθόδους hacking που χρησιμοποιεί η ΑΕΕ. Ποιος είναι υπέρ της πρότασης. Ποιος είναι κατά. Αποχές. Η πρόταση απορρίπτεται. Επομένως, η ημερήσια διάταξη παραμένει ως έχει. Ο κύριος Βίμπερτ, διαδικαστικό. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα καταρχήν να μην γίνει η ψηφοφορία που έχουμε αύριο για τα όπλα, γιατί η οδηγία αυτή δεν έχει την επιπτωσιολογική μελέτη που είχαμε ζητήσει, άρα λοιπόν δεν θα έπρεπε να την ψηφίσουμε. Θα ήθελα λοιπόν να διαγραφεί το σημείο αυτό για τα όπλα και την οπλοκατοχή από την ημερήσια διάταξη μέχρι να μας παρουσιάσει τη μελέτη αυτή η Κομισιόν. Ο κύριος Νόστοκ. πριν μιλήσω καν, περιμένετε λίγο και αρχίζετε μετά τη Γιούχα. Κοιτάξτε, πέμπτη βράδυ έγινε το αίτημα και παρακαλώ να αναφέρετε τον τίτλο και όχι μόνο το έγγραφο. Αφορά τη συνεργασία μεταξύ διακινητών και ΜΚΟ που κάνουν ε, υποτιθέμενες δράσεις ε, διάσωσης. Είναι κομμάτι της παράνομης διακίνησης στη Μεσόγειο και παρακαλώ να μπει ο τίτλος όπως συνηθίζεται και όχι μόνο ο αριθμός του εγγράφου. Απαντήσω στην κυρία Νόρστοκ. Η απόφαση του τίτλου ε, γίνεται από τη διάσκεψη των Προέδρων και ο Πρόεδρος συμμετείχε σε όλες τις συνεδριάσεις. Γνωρίζετε πάρα πολύ καλά λοιπόν περί τίνες πρόκειται. Κυρία Βίμπερκ, υπάρχουν ε, ε, προθεσμίες για να ζητήσετε αλλαγές και είστε εκτός προθεσμιών. Τρίτη, η ομάδα της GUNGL ε, ζήτησε μια δήλωση της Αντιπροέδρου ε, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής υπάτης εκπροσώπου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις εξωτερικές υποθέσεις ε, και την πολιτική ασφαλείας για τις κατεδαφίσεις κατοικιών και δομών που ανήκουν σε Παλαιστινίου να προσθεθεί ως τρίτο θέμα το απόγευμα μετά τη δήλωση της υπάτης εκπροσώπου για τις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το ο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των ΗΠΑ Εθνών του 2017. Η συζήτηση θα ολοκληρωθεί με ψήφισμα. Να δώσω το λόγο στον κύριο Σιλικιώτη για να μας παρουσιάσει το αίτημα της ομάδας του. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, η εκκληματική πολιτική των κατεδαφίσεων που εφαρμόζει το Ισραήλ σε βάρος του Παλαιστινιακού λαού συνεχίζεται. Χθε ήταν η τελευταία ημέρα διορία που δόθηκε από τι Ισραηλινέ Αρχέ στην κοινότητα των Βεδουίνων και να κατεδαφίσουν τα σπίτια του στο χωριό Καν Αλάχμα στη δυτική όχθη τη Παλαιστίνη. Η κοινότητα αυτή των Βερτιουίνων κινδυνεύει άμεσα, αποτελείται από 140 κατοίκου, εκ των οποίων τα περισσότερα είναι παιδιά. Μάλιστα, να σα πω ότι στον οικισμό ανεγέρθηκε νηπιαγωγείο με χρηματοδότηση τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Η αντιπροσωπεία του Ευρωκοινοβουλίου με την Παλαιστίνη είχαμε επισκεφτεί πρόσφατα αυτό το χωριό και λόγω της παρουσίας μας εκεί οι ισραηλινές αρχές έχουν αναβάλει την κατεδάφιση η οποία είχε προγραμματιστεί να γίνει τον φεβρουάριο. πρέπει να πω ότι με βάση στοιχεία του οηε το 2016 έγιναν οι πιο πολλές κατεδαφίσεις από το ισραήλ το 2017 οι ισραηλινές αρχές έχουν ήδη κατεδαφίσει 172 παλαιστινιακές ζωνές στην περιοχή γάμα και στην ανατολική ιερουσαλήμ. είναι μια πολιτική αυτή του ισραήλ να κατεδαφίσουν τους οικισμούς να επεκτείνουν τους παράνομους επικισμούς των ισραηλινών και να χωρίσουν τη δυτική όχθη στα δύο. είναι ώρα η ευρωπαϊκή ένωση να δράσει άμεσα να διασφαλίσει ότι οι παράνομε κατεδαφίσει και οι παράνομε επεκτάσει στον ισραηλινό οικισμό θα τερματιστούν. το ευρωπαϊκό κοινοβούλιο πρέπει να στείλει το μήνυμα αντιτίθεται σε αυτέ τι παράνομε κατεδαφίσει αντιτίθεται στι παράνομε επεκτάσει των ισραηλινών οικισμών και στηρίζει τη λύση δύο κρατών η οποία είναι η μόνη επιλογή σήμερα για να επικρατήσει μόνιμη ειρήνη ε, στην ευρύτερη μέση ανατολή. ευχαριστώ πρόεδρε. Υπάρχει κάποιος ο οποίος θα ήθελε να παρέμβει κατά της πρότασης ε, της ομάδος ε, GUNGL. Παρακαλώ. Monsieur le Président. Κύριε Πρόεδρε, είμαστε κατά αυτής της πρότασης. Γιατί ξέρετε πως στην κοινότητα Κάνα Λαχμέρ που είναι στην ε, ζώνη αυτή, το παράνομο είναι ακριβώς αυτές οι κατασκευές που βρίσκονται στην ε, περιοχή γιατί βρίσκεται υπό, Ισραηλινή, ε, υπό Ισραηλινικό έλεγχο όλη αυτή η περιοχή και οι Παλαιστίνοι δεν ζήτησαν έγκριση για να χτίσουν και νομίζω ότι οι δικές τους κατασκευές που αναφέρατε εσείς είναι παράνομες. Και εφόσον δεν έχουν εξαντλήσει κάθε νόμιμη διαδικασία, νομίζω ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος εμείς να σπείρουμε τη σύγχυση με τον τρόπο με τον οποίο προτείνει ο συνάδελφος, ο οποίος μίλησε δε ε, και για τις επικείμενες ε, ε, προσπάθειες που θα γίνουν για να αποπακρινθούν τα κτίρια αυτά. Ε, είμαστε ακόμα στο Μάρτιο, οπότε δεν νομίζω ότι υπάρχει πρόβλημα. Allora, pongo ora in votazione. Ωραία. Θα ψηφίσουμε με ονομαστική κλίση το αίτημα της GUNGL για να προσθεθεί στη συζήτηση της Τρίτης μετά από τη δήλωση της Αντιπρόεδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Υπάτη εκπροσώπη για τι προτεραιότητε της Ένωσης ε, για το ε, Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών και τη συνεδριάση του 2017, μια δεύτερη δήλωση για τις κατεδαφίσεις ε, κατοικιών και κατασκευών που ανήκουν σε Παλαιστινίους. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση τη ψηφοφορίας. Η πρόταση απορρίπτεται. Η ημερήσια διάταξη λοιπόν παραμένει ως έχει. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να μιλήσω για την Τουρκία και τις δηλώσεις του κυρίου Ερντογάν, ο οποίος τοποθετείται κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και είδαμε τις ε, δηλώσεις ε, του κυρίου Ερντογάν που αποκαλεί τους Ολλανδούς Λίδιν φασίστες ε, και ναζί. Δεν είναι δυνατόν, δεν μπορούμε να το ανεχτούμε ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Πρέπει να προσθεθεί στην ημερήσια διάταξη αυτής της εβδομάδας. Ξέρω ότι έχει προγραμματιστεί για τον Απρίλιο, αλλά δεν είναι δυνατόν να κρυβόμαστε πίσω από τις ε, διαδικασίες. Πράγματι, ομολογώ, είμαι εκτός της ε, προθεσμίας, αλλά μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Να συζητήσουμε αυτό το οποίο είναι πραγματική επίκαιρη πολιτική, σαν πραγματική πολιτική σε ένα πραγματικό κοινοβούλιο και να γίνει μια συζήτηση για την Τουρκία. Οι κανόνε πρέπει να γίνονται σεβαστοί. Ο κύριο Βιευσκόφσκι. Ευχαριστώ πολύ. Νομίζω πως ο τρόπος που διαχειρίζεστε τη συνεδρία είναι εξαιρετικά λογικός και βεβαίως σεβόμαι και τον τρόπο με τον οποίο δίνετε το λόγο στους συναδέλφους. Αλλά μην ξεχνάτε το άρθρο 184. Δηλαδή, εάν κάποιος ε, βουλευτής θέλει να καταθέσει τέτοια δήλωση ή να κάνει τέτοια δήλωση, νομίζω ότι θα πρέπει να το κάνει στα πλαίσια του, ε, της παρέμβασης του ενό λεπτού, όπως κάνουμε όλοι οι υπόλοιποι. Οπότε νομίζω ότι ο συνάδελφος θα έπρεπε να ακολουθήσει το άρθρο 184 και τα όσα εκεί θεσπίζονται. Έτσι είναι ο σωστός τρόπος για να προχωρήσουμε. Και εκεί μπορεί να κάνει όσα σχόλια επιθυμεί. Σας ευχαριστώ πολύ για τη συμβουλή σας. Και τώρα, παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, κάτι για την ημερήσια διάταξη. Θα ήθελα να υπενθυμίσω πως ε, υπάρχει ένα εναλλακτικό ψήφισμα που κατέθεσε ο κύριος ε, Νταντών σε σχέση με την έκθεση ίδιας πρωτοβουλίας για τα για τα πειραματόζωα, ε, κάτι το οποίο παραβιάζει το άρθρο 170 παραγραφός 1 του κανονισμού. Τώρα μάλιστα διαπιστώνω πως μετά την ε, εκπνοή της ε, προθεσμίας το κείμενο περιεκοπεί. Αν ο λόγος ήταν ένα τεχνικό πρόβλημα, όπως αναφέρεται στο άρθρο 117 παραγραφός 4, μπορούν ε, κατ' εξαίρεση μετά τη λήξη της προθεσμίας με τη σύμφωνη γνώμη του Προέδρου να αλλάξουν οι προτάσεις εάν πρόκειται για συμβαστικές ε, τροπολογίες ε, ή για τεχνικό λάθος. Κάτι το οποίο όμως σημαίνει ότι θα πρέπει να ζητηθεί η σύμφωνη γνώμη του Κοινοβουλίου πριν από την ψηφοφορία. Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα λοιπόν να σας ρωτήσω εάν εσείς θεωρείτε ότι επιτρέπεται η κατάσταση του εναλλακτικού ψηφίσματος ε, του ΕΛΚ ή αν θα τεθεί σε ψηφοφορία όπως ορίζει ο κανονισμός. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Allora... Η πρόταση του ΕΛΚ ήταν πιο μακροσκελή από ό,τι επιτρέπεται, διότι όπως γνωρίζετε η εναλλακτική πρόταση πρέπει να είναι πιο σύντομη από την αρχική πρόταση. Οι υπηρεσίες μας όμως, όπως ε, γίνεται πάντα, ενημέρωσαν το ΕΛΚ και το κείμενο ε, περιορίστηκε. Επομένως, επειδή ακριβώς ε, πρόκειται μόνο για ένα τεχνικό πρόβλημα που αφορούσε ε, το μήκος του κειμένου και όχι ε, το περιεχόμενο και την ουσία, θεωρώ ότι γίνεται παραδεκτό αυτό το έγγραφο. Επαναλαμβάνω, πρόκειται απλώς για ένα τεχνικό πρόβλημα το οποίο επέλυσαν οι δύο υπηρεσίες του Κοινοβουλίου. Σας ευχαριστώ. Να δώσουμε αμέσως τώρα το λόγο στον κύριο Εκ, ο οποίος είναι εισηγητής για την έκθεση για τον Ιδράγυρο.